Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην απόψινή συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Κέβεν Κάντιφ που έχει οριστεί ως υποψήφιος από τις Ιρλανδικές Αρχές για να γίνει μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως και άλλοι υποψήφοι τους οποίους ακούσαμε νωρίς το πρωί, υπό την ίδια διαδικασία, ο υποψήφιος μιλά για πέντε λεφτά και έπειτα ο εισηγητής κάνει μια πρώτη εισήγηση και μετά δίνει παίρνει το λόγο τα μαλλιά. Συμφωνείτε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Σας προτείνω να δώσουμε το λόγο αμέσως στον κύριο Κάρντιφ για πέντε λεπτά και για ολόκληρη τη διαδικασία έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε λέγομαι Kevin Cardiff, είμαι υποψήφιος της Ιλλανδικής Κυβέρνησης για τη θέση του μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιόν σας και να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Νομίζω είναι η πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη και εργασία που έχω χρειαστεί να περάσω. Έχετε το βιογραφικό μου, γι' αυτό θα σταθώ μονάχα σύντομα στα θέματα αυτά. Τελείωσε το 1979 το γυμνάσιο, το Λύκειο μάλλον. Έκανα το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ με μια αθλητική υποτροφία και αποφύτησα το 1983 με πτυχίο σε Ιστορία και Ψυχολογία συνέχισε στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Δουβλίνου για μάστερς για... και μετά μπήκα στις, ε, στη δημόσια υπηρεσία της Ιρλανδίας για θέματα ισότητος. Έχω μία πορεία στις, στο δημόσιο τομέα, καταρχήν σε σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις χρηματοοικονομικές αγορές, ήταν η μία πτυχή η δεύτερη πτυχή ήταν οργανωτικά θέματα και θέματα ανθρωπίνων πόρων. Άρχισα να εργάζομαι σε εργασιακά θέματα και σε συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Μετά πέρασα σε θέματα όπως ελευθερία πληροφόρησης, έλεγχος διοικητικών δαπανών. Και μια τρίτη πτυχή αυτής της καριέρας μου ήταν όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσω θέματα φορολογικής πολιτικής και εκεί προείδρευσα στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης φορολογικών ε, δαπανών, κάτι το οποίο πιστεύω ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με την εργασία του ελεκτικού συνεδρίου. Το φθινόπωρο του 2008 ήμουν υπεύθυνο για το τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και φορολογικών θεμάτων και στη συνέχεια ο Υπουργό και ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μου ζήτησαν να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και αυτό έπραξα μέχρι ότου διορίστηκα το Φεβρουάριο του 2010 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Θα ξέρετε ότι το σύστημα του Ιρλανδικού, <clears throat> της Ιρλανδικής κυβέρνησης σύνολο έχει να αντιμετωπίσει μια τεράστια μάχη στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και τον έλεγχο των οικονομικών ενώπιον μιας μεγάλης κρίσης. Βρέθηκα στο μάτι, στον πυρήνα της ε, διαδικασίας αυτής σε πολλούς τομείς και νομίζω ότι οι προτάσεις μου και οι εισηγήσεις μου έχουν γίνει θετικά δεκτές από την κυβέρνηση και από άλλους φορείς. Η Ιρλανδία έχει χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει τα θέματα της κρίσης και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι για κάθε ένα από τους τομείς κρίσης, χρηματοπιστωτικός τομέας, οικονομία, δημοσιονομία. η Ιρλανδία είναι πια στο δρόμο της επιστροφής σε μια ομαλή κατάσταση και η σωστή απόδοση της χώρας μας είναι δείγμα της αποφασιστικότητας των Ιρλανδών πολιτών να ξεπεράσουν την κρίση αυτή. Όταν ο Τίσοκ, ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, μου ζήτησε να γίνω υποψήφιος για το ελεκτικό συνέδριο, θεωρώ ότι είναι μια τιμή προς εμένα προσωπικά, αλλά και μία τιμή για το φορέα στον οποίο εργάζομαι. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να συμβάλλω στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί μπορώ να φέρω την εμπειρία μου λόγω της καριέρας μου στο δημόσιο τομέα, αλλά και επίσης χάρη και στα τρία ή τέσσερα χρόνια που έχω εργαστεί κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Μια δύσκολη αλλά πάρα πολύ παιδαγωγική εμπειρία. Η Ευρώπη πολυ δυσκολε συνθηκες μια δυσκολη αλλα παρα όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες και ενδεχομένως η Ιρλανδία θα μπορέσει αρνητικά ίσως ή λιγότερο θετικά να δώσει τα πορίσματα της εμπειρίας της τα τελευταία χρόνια και θα είμαι πάρα πολύ διαθέσιμος να χρησιμοποιήσω αυτή την εμπειρία που απέκτησα στο ελεκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και στη συνέχεια ο εισηγητή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάρτιφ για την παρουσίασή του. Διαβάσαμε προσεκτικά και το βιογραφικό του. Φαίνεται ο κύριος Κάρντιφ να είναι ένας δημόσιος αξιωματούχος ο οποίος κράτησε υψηλά αξιώματα, χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις και έχει βοηθήσει την κυβέρνησή του σε συνθήκες κρίσης. Έχουμε λοιπόν σημεία τα οποία δείχνουν και την προσωπική σας αξία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Κάρντιφ οι συνάδελφοί μου ενδιαφέρονται κυρίως για δύο θέματα. Μέσα στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής κρίσης την οποία αναφέρθηκατε στην Ιρλανδία, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είδους αλυσίδα διοίκηση, κατά κάποιο τρόπο, τι είδους πυραμίδα εξουσίας υπήρξε στην Ιρλανδία για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, ώστε να υπάρχει πολιτική εποπτεία και όχι απλώς σε επίπεδο διοικητικό επίπεδο και θα ήταν χρήσιμο να μπορέσετε να μας εξηγήσετε με περισσότερες λεπτομέρειες πώς ακριβώς λειτουργήσε αυτό το σύστημα στην Ιρλανδία και πώς υπήρξε λογοδοσία ενώπιον του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στον τομέα αυτό και θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό ήσασταν υπεύθυνο για αυτές τις εκθέσεις. Ένα άλλο δεύτερο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί και αυτό προέρχεται από τις προηγούμενες μέρες λίγο πριν από τη σημερινή ακρόαση. Είναι μια κατάσταση φαινομενικής τουλάχιστον διπλής λογιστικής για δύο φορείς που ήταν υπεύθυνοι για το Ιρλανδικό χρέος. Φαίνεται ότι υπήρξε μια αλλαγή σε σχέση με τους φορείς που έπρεπε να κάνουν την επαλήθευση του χρέους και για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρξε διπλή λογιστική και διπλή απεικόνηση του ίδιου αυτού χρέους. Λαθασμένη κατά συνέπεια καταγραφή. Και υπήρξε μια διαμάχη για το θέμα αυτό. Εσείς προφανώς θα πρέπει να είσαστε ενήμερος για τα θέματα αυτά και θα ήθελα να ξέρω ποια ήταν η δική σας εικόνα για τα σφάλματα τα οποία υπήρξανε κατά πόσο εσείς εμφανιστήκατε εναντίον των πολιτικών υπευθύνων, δηλαδή στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο για να εξηγήσετε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε αυτή την ευθύνη, την ευκαιρία να μας εξηγήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δική σας προσωπική εμπλοκή σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Cardiff, you have the floor. Thank you. Κύριε ευχαριστώ πρόεδρε. σε ό,τι αφορά την ανάμειξή μου στα τραπεζικά ζητήματα, η υποψηφιότητά μου είναι κάπως αμφιλεγόμενη στην Ιρλανδία. Όσοι με γνωρίζουν και γνωρίζουν ε, το έργο μου, ε, με σέβονται. Η συμβολή μου, ε, η μου εκτιμάται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τραπεζική κρίση και το ποιος ήταν υπεύθυνος γιατί. Στην Ιρλανδία εστιαστήκαμε κυρίως στο Σεπτέμβριο του 2008, όταν η κρίση χτύπησε και σημείωσε μια κρίση τουλάχιστον στη φαντασία του κοινού. Τότε ήμουν ε, ο επικεφαλής του τμήματος ε, για θέματα ε, τραπεζών στο Υπουργείο Οικονομικών και προφανώς υπέβαλα εκθέσεις στον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό. Στην Ιρλανδία τέθηκε το θέμα των τραπεζικών εγγύσεων. Εγώ ήμουν σύμβουλος της κυβέρνησης εκείνο το απόγευμα μαζί με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών και τον ε, Υφυπουργό και με συμβούλους όπως τον ε, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, το Γενικό Εισαγγελέα και το καθεξής και ενεργά συμμετείχα στην συζήτηση εκείνη. Επεσήμενα αυτά που ήθελα να επισημάνω για να ξέρει η κυβέρνηση ποια ήταν η θέση μου. Και νομίζω ότι ήταν ένα θέμα που πέρα από τις θεσμικές, αν θέλετε, ε, διαπιστώσεις προβαίνει κανείς και σε προσωπικές ε, τοποθετήσεις. δεν περιορίζεται κανείς μόνο στην θεσμική γραμμή. Όταν αντιμετωπίζει κανείς μια πραγματική κρίση, τα άτομα, οι προσωπικότητες πρέπει να τοποθετούνται και αυτό το έπραξα. Αλλά ήμουνα υπεύθυνο και για μεγάλο τμήμα της προπαρασκευής, της προετοιμασίας για την κρίση. Εγώ και η ομάδα μου λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να προετοιμάσουμε όχι ένα, αλλά δύο, ίσως και τρία νομοθετήματα για την αντίδραση στην κρίση. Και είχαμε διάφορα νομοθετήματα στο γραφείο μας. Σχέδια για την ανάληψη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για εγγυήσεις, για swaps τύπου Ηνωμένου Βασιλείου. Όταν σημειώθηκε λοιπόν η κρίση, όταν ξέσπασε η κρίση, η κυβέρνηση είχε διάφορες ε, επιλογές. Αυτή ήταν η δουλειά μου, να διασφαλίσω ότι είχαν επιλογές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ε, κατεπήγον χαρακτήρας και ασφαλώς και καλό θα ήταν να είχαμε πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αλλά από την άλλη ξέρω ότι εντός εβδομάδες είχε σημειωθεί η πτώση της Lehman Brothers στην Αμερική και ακολούθησαν τα υπόλοιπα γεγονότα στην Ευρώπη. Νομίζω την ίδια ημέρα. RBS στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπήρχε περιθώριο στην ε, περίσταση αυτή να κινηθούμε πιο αργά. Εκείνο το απόγευμα, ωστόσο, η συζήτηση ήταν αρκετά ψύχρεμη σε σχέση με τις ε, δυνατότητες που υπήρχαν. Η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό τελικά έλαβαν τις αποφάσεις και όπως είπα και δημόσια, στο Ατλαντικό σύστημα υπήρξε κριτική κατά των πολιτικών των υπουργών. Αλλά δήλωσα δημόσια ότι στην φάση εκείνη υπήρχε κίνδυνος οι πολίτες να μην έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους την επόμενη εβδομάδα. Άρα θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι αποφάσεις ε, που ελήφθησαν δημιούργησαν ε, ένα περιθώριο, ένα χρονικό περιθώριο και προστάτευσαν τους πολίτες μας και πολίτες ε, σε άλλα τμήματα της Ευρώπης από τον κίνδυνο επιμόλυνσης και μια άμεση καταστροφή στο σύστημα διπλής καταγραφής, διπλής καταμέτρησης. Είναι λίγο διαφορετικό και σε αυτό το σύνδημα είμαι ο επικεφαλής για τις διοικητικές αποφάσεις. Όχι απόλυτα, γιατί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ε, μπλέκεται επίσης. Αλλά έπρεπε ως ε, υπεύθυνο αξιωματούχος να πω ότι ήταν δική μου ευθύνη και ευθύνη του δικού μου τμήματος. Πρέπει να είμαι προσεκτικός γιατί μπορεί να είναι κάποιοι Ιρλανδοί οι οποίοι με ακούν αυτή τη στιγμή. Δεν χάσαμε τα λεφτά κανένας. Δεν εξαφανίστηκαν τα λεφτά αυτά. Πρέπει να το ξέρουν όλοι οι Ιρλανδοί πολίτε Δεν έχουν χαθεί χρήματα από τις τράπεζες. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι μία καταγραφή μίας συναλλαγή έγινε σε δύο βάσεις. Η, ένα δάνειο της ε, χρηματοπιστωτικής μας υπηρεσίας εμφανίστηκε σαν να έχει γίνει κατευθείαν από την αγορά ενώ έγινε στην πραγματικότητα από το Εθνικό θησαυροφυλάκιο και δεν έγινε σωστή αναφορά για τα θέματα αυτά που οδήγησε σε διπλή καταμέτρηση, σε δύο λαθασμένες, σε δύο εγγραφές. Εγώ το κατανόησα αυτό μετά από λίγες ώρες από τη στιγμή που έγινε γνωστό το θέμα αυτό στο ευρύ κοινό και από τη στιγμή που έγινε αυτό φυσικά γνωστό στον αρμόδιο υπουργό, το δημοσιοποίησε όπως ήταν το καθήκον του μάλλον πριν το μάθει το κοινό και το δημοσιοποίησε ο Υπουργό όπω ήταν το καθήκον του και περάσαμε στη συνέχεια σε μια διαδικασία ελέγχου σε εσωτερικό επίπεδο και υπάρχει και μια, ένας ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος για το συνολικό σύστημα του Υπουργείου μας. Αλλά αυτό μπορεί να κάνει μονάχα κανεί όταν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πηγαίνουμε σε μια επιτροπή και λέμε ναι βεβαίως κάνουμε ένα έλεγχο να δούμε τι έγινε. Αλλά Αυτά πρέπει να γίνονται. Όταν συμβαίνει ένα τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει να προσπαθήσει κανεί να το επιλύσει. Στην αρχή πρέπει να δώσει μια γρήγορη απάντηση και μετά να δει τι αιτίε αυτού του προβλήματο. Και από τη δική μου άποψη, εγώ είμαι ικανοποιημένο γιατί δεν θα επαναληφθεί αυτό το σφάλμα. Αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν σφάλματα. Εγώ ω υπεύθυνο του λογιστικού τμήματο έχω την υπευθυνότητα να ασχολούμαι με αυτά τα πιθανά σφάλματα. Μπορείτε να ρωτήσετε πού ακριβώ προέκυψε αυτό Ίσως κάποια άτομα εδώ πέρα διακυβεύεται η φήμη τους, η καριέρα τους. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένους πιθανούς υπεύθυνου. Δεν θα ήταν δίκιο για μένα να πω ότι φταίει η τάδε ή η δίνα υπηρεσία. Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η... ο έλεγχος αυτός και η επισκόπηση της κατάστασης για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευχαριστώ. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο στα μέλη μας, τα οποία θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα η Ίγκεμπορκ Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάντεφ, βλέπω ότι έχετε ένα ισχυρό λόμπι που σας υποστηρίζει. Μας στείλανε πολλά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, δεν τα έχω φέρει όλα αυτά στην αίθουσα από μένα, αλλά εντυπωσιάζομαι που τόσοι πολίτες μιας ε, χώρας μέλους απευθύνθηκαν σε εμά και είπανε κάντε ό,τι μπορείτε για να μην ε, γίνει μέλος του ελεκτικού συνεδρίου ο κύριος Κάντιφ. Τι θα πούμε στους πολίτες λοιπόν αν σας εγκρίνουμε. Δεύτερο, θα ήθελα να μας πείτε ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου τι μπορείτε να μας πείτε ότι έχουμε μάθει από την κρίση αυτή, από τη χώρα σας. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Σημείο 3 σε σχέση με τα προσόντα σας. Πρέπει να πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της Ιλλανδίας ουσιαστικά τιμωρήθηκε από τους πολίτες έχασε τις εκλογές. Και υπάρχει και μια έκθεση του Independent ε, Review Panel που τη γνωρίζετε πολύ καλά και δίνει 50 συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοοικονομική κρίση θα έπρεπε να είχε τύχει διαχείρισης στην Ιρλανδία και κάποιες από αυτές τις συστάσεις αφορούν και το δικό σας λειτουργήμα. Θα ήθελα λοιπόν σε σχέση με αυτό να ξέρω ποια είναι η θέση σας για το σύνολο αυτό των συστάσεων. Αν πράγματι συμφωνείτε και εσείς ότι μπορεί κανείς να συναγάγει ότι υπήρξε μια συνολική οργανωτική αποτυχία στον τομέα αυτό στην Ιρλανδία. Φυσικά είσαστε ένα πάρα πολύ σημαντικός υποψήφιος γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος διασώσεως που πληρώνει για, το, για τα σφάλματα της Ιρλανδίας στο παρελθόν. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να υπάρξει και μεγαλύτερη υπευθυνοποίηση για τα θέματα αυτά. Μπορεί κανείς να συναγάγει ότι υπήρξε λοιπόν μια οργανωτική αποτυχία συνολικά στην Ιρλανδία. Ο κ. Κάντεφ να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Κρέσλε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξαν πολλά ηλεκτρονικά γράμματα προς εσάς και τι να σας πω με εκπλήσει. Δεν πάω και για εκλογές. Δεν πάω και για πρωθυπουργό. Φαντάζομαι ότι τέτοια πίεση δέχεστε συνέχεια βέβαια εσείς. Μπορώ να την εξηγήσω μόνο λέγοντας ότι στην παρούσα φάση είναι τεράστια η αγανάκτηση και πολύ φυσική στην Ιρλανδία για την κρίση που διερχόμαστε. Υπάρχει μεγάλη αποφασιστικότητα στην Ιρλανδία να την αντιμετωπίσουμε την κρίση, αλλά ασφαλώς και να ανακτήσουν ο κόσμος με το γεγονός ότι αναγκάζεται να, να κάνει αυτά που κάνει. Και στην παρούσα φάση να σας πω ότι δεν έχουν μείνει και πολλοί αξιωματούχοι που ήταν ε, και συμμετείχαν στην όλη διαδικασία τότε. Άρα, ε, ανακύπτει ερώτημα του γιατί έχω μείνει εγώ. Δουλεύω κάθε μέρα και δουλεύω όσο καλύτερα μπορώ με το αίσθημα ευθύνη που έχω. Δεν έχω την αίσθηση ότι απογοήτευσα κανέναν ποτέ, γιατί έκανα πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Αλλά αυτό ίσως να μην αρκεί. Και νομίζω ότι χρειάζονται κάποια εξωτερικά αποδεκτικά στοιχεία. Τα μοναδικά αποδεκτικά στοιχεία τα οποία έχω να προσκομίσω πέρα από την παρουσίασή μου εδώ και την παρουσία μου εδώ είναι ότι ήμουν γενικός γραμματέας ε, του ε, Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το 2010. Όταν άνοιξε μία θέση λοιπόν και χρειάστηκε κάποιος να αντιμετωπίσει την τεράστια πίεση στην οποία εφιστάμεθα, η κυβέρνηση αποφάσισε τότε να με διορίσει. Ήξεραν καλά τη δουλειά μου μέχρι τότε και είχαν ε, την ευκαιρία να διαλέξουν κάποιον άλλον, αν ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσα να τα απεξέλθω. Όταν ασφαλώς ε, σχηματίζεται μια νέα κυβέρνηση, πάντα υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση αξιωματούχων. Παρ' όλα αυτά, και η νέα κυβέρνηση, μετά από αναδιοργάνωση του τμήματό μου, με έβαλε στη θέση αυτή. Εργαζόμουν για κάποιους μήνες μάλιστα και για δύο υπουργεία, το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο, πρέπει να ομολογήσω και ήμουν ουσιαστικά, αν θέλετε, το άτομο το οποίο έπρεπε να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει συνέχεια. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μετάβαση σε μια νέα κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, τα διάφορα προγράμματα. Και τώρα η κυβέρνηση με προτείνει ε, ως υποψήφιο για το ελεκτικό συνέδριο. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την σημερινή κυβέρνηση είναι κάτι, απασχολείται μάλλον και ασχολείται με κάτι που μας το ανακοινώνει κάθε μέρα. Να συμβάλλει η Ιρλανδία πιο καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θεωρώ ότι θα με πρότειναν για τη θέση αυτή αν είχαν την αίσθηση ότι δεν θα τους εκπροσωπούσα σωστά, ότι δεν θα εκπροσωπούσα την χώρα σωστά. Δεν έχω κάποιο έλεγχο να σας δείξω πόσο καλά τα πήγα, αλλά νομίζω ότι γενικά ο κόσμο έχει την ευκαιρία να με αξιολογήσει και μάλιστα με θετικό τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έκανα τεράστια ασφάλματα, γιατί σε μια τέτοια περίοδο κρίση ε, διαπράττει κανεί τεράστια ασφάλματα σε κάποιε περιπτώσει. Και έχω πραγματικά και πολλού σπουδαίους συναδέλφου που έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τα διδάγματα που αντλήσαμε. Είναι πολλαπλά. Αλλά αν έκανα λάθη και έχω παραδεχτεί κάμπος από αυτά. Θα έλεγα ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε αρκετά γρήγορα την κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις. Πάντα υπάρχει λόγος να μην αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση και συνήθως είναι και πολύ λογικός και πολύ θεμητός ο λόγος αυτός. Όταν ε, ξεκινά κανείς να δουλεύει με πολύ δημόσιο τρόπο, αυτό συνήθως επιταχύνει την κρίση. Αν ε, προσθέσει προσωπικό σε κάποιον τομέα, θα το προσέξει ο κόσμο ότι προετοιμαζόμαστε για την κρίση και έτσι θα επιδεινώσει την κατάσταση αυτά από μόνο του. Κάτι σημαντικό στην Ιρλανδία. Προσπαθούμε να ελαφρώσουμε τον ε, δημόσιο τομέα μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση με λιγότερο προσωπικό αλλά σε κάποιε περιπτώσει πολύ απλά πρέπει να αντιληφθεί κανεί το μέγεθο τη κρίση και να αναλάβει τους κινδύνους και να κινηθεί γρήγορα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα και το δίδαγμα που αντλώ για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ιρλανδία, σε ό,τι αφορά την έκθεση. Right. Ανατέθηκε στην οργάνωση του Υπουργείου των Οικονομικών πριν λίγες εβδομάδες ε, αφότου ε, διορίστηκα Γενικός Γραμματέας και την ξεκίνησα εγώ κατόπιν εντολής του Υπουργού. Νομίζω περιλαμβάνει 50 συστάσεις, ε, αλλά απογοτευτήκαμε. γιατί σκοπός ήταν να μάθουμε από αυτά που είχαμε περάσει και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο Υπουργείο Οικονομικών για το μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και έχω έξι άτομα που 7-8 που έχουν ζητήσει το λόγο για να θέσουν ερωτήσεις. Οκτώ άτομα, οκτώ άτομα. Θα δώσω το λόγο σε αυτούς που ζήτησαν το λόγο, σε ομάδες των τριών. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάρντιφ να απαντήσει σε τρία λεπτά. Ελπίζω να έχετε όλη την ευκαιρία να μιλήσετε. Κύριε Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λεπτά. Κύριε Κάρτιφ, ε, θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε. Να τη διατυπώσω με άλλα λόγια. Θεωρείτε ότι υπάρχει θεσμική προσωπική ε, ευθύνη σας για την Ιρλανδική τραπεζική κρίση. Δεύτερη ε, ερώτηση. Η υπόθεση που έχουμε μπροστά μας, μιλάτε σε ό,τι αφορά την απάντηση στις ερωτήσεις της εισηγητριάς. Μιλάτε για ακρόαση στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις που διαβάσαμε στον τύπο, θεωρείτε ότι εμπίπτουν στο πεδίο της προσωπικής σας ευθύνης για την τραπεζική κρίση. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τσάλντερς. Η κυρία, διορθώνει ο πρόεδρος, συγγνώμη. Yes, um, I would like to ask... Ναι, θα ήθελα να θέσω δύο ε, ερωτήσεις. Πείτε μου, κύριε Κάρτιφ, γιατί θεωρείτε ότι σας ε, προτείνουν για τη δουλειά αυτή. Και δεύτερη ερώτηση. Τι θεωρείτε ότι περιλαμβάνει αυτή η θέση εργασίας. Ε, θεωρείτε ότι είναι εύκολο, δύσκολο το έργο αυτό. Σημαίνει ότι είναι ε, κάτι το πανεύκολο. Πείτε μας ε, πώς βλέπετε τη δουλειά αυτή για την οποία σα προτείνουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σούντεργκάρντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ τι ρετήσει έχω να κάνω. Πρώτη. Είδατε ότι από τον Αύγουστο του 2010 έγιναν τρεις φορές λάθη στην αλυσίδα εντολών, όπου δεν, έ δεν λάβατε εσείς τις απαραίτητες πληροφορίες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες σας, κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι κάναν λάθη ή έχει να κάνει αυτό με μια εσφαλμένη νοοτροπία στα θεσμικά όργανα, τα οποία έπαιξαν τόσο κεντρικό ρόλο. Δεύτερη ερώτηση. Που προκύπτει από αυτά που μας θέσατε και μας παρουσιάσατε εσείς. Είπατε ότι ε, σημειώθηκε η καταστροφή της Lehman Brothers. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν ήταν φυσική καταστροφή, ήταν κάτι το οποίο μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει εκ των προτέρων. Γιατί η κρίση ήταν επικείμενη. Είναι κεντρική η θέση σας, ήταν κεντρική η θέση σας στο Υπουργείο Οικονομικών το 2006 Πώς μπορείτε να περιγράψετε το υπόβαθρο της κρίσης στην Ιρλανδία. Κατανοώ την καλή δουλειά που έγινε όταν ξέσπασε η κρίση, αλλά πριν ξεσπάσει η κρίση υπήρχαν διάφορες ενδείξεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Προφανώς αυτό δημιουργήσε κάποια, κάποια σκέψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι σκέψεις είχαν γίνει λοιπόν τότε μεταξύ του 2006 και του πραγματικού ξεσπάσματος της κρίσης. Πείτε μας δύο λόγια. Ο κ. Κάρντιφ έχει το λόγο για να απαντήσει σε τρία λεπτά. Το έχω περάσει όλο αυτό το... Τα θέματα έχω σκεφτεί στο μυαλό μου και νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω μια συνεκτική απάντηση. Ό,τι αφορά την δακτυλοδειξία και την μεταφορά του φτεξίματος. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνει κανείς. Η κρίση τραπεζική και η κρίση της ελληνικής οικονομίας ήταν το αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικών σχεδίασης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατά κύριο λόγο. Δεύτερον, από έλλειψη κατανόησης και σωστής εποπτείας στο ρυθμιστικό σύστημα το οποίο έπρεπε να ελέγχει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τρίτον για είναι αποτέλεσμα του τρόπου διαχείρισης του προβλήματος όταν εξελιχθήκε η κρίση και της έλλειψης κατανόησης της κλίμακος αυτού του προβλήματος. Εγώ δεν ήμουν κομμάτι του ρυθμιστικού συστήματος, δεν ήμουνα στο, στο Συμβούλιο Ρυθμιστών της Κεντρικής Τράπεζας. Το πρώτο τμήμα της δεκαετίας 2000 ήμουνα μεταξύ αυτών οι οποίοι θέσπισαν τους κανονισμούς για τη δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά οι εκθέσεις για την κρίση που ανέφεραν ποιες ήταν οι δυνατότητες μέσα σε αυτή την ρυθμιστική δομή δεν χρησιμοποιηθήκανε στην συνέχεια και δεν χρησιμοποιήθηκε επαρκώς η νομοθετική οδός ρύθμισης. Σε ό,τι αφορά την κατανόηση της κρίσης εν τη της, πρέπει να πω ότι πράγματι δεν κατανοήσαμε εν την τεράστια, την τεράστια διάσταση αυτής της κρίσης στις ε, υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ακόμα και το Σεπτέμβριο του 2008 δεν ήταν ακόμα ορατές οι απώλειες που θα επακολουθούσαν. Και για μένα και για πολλούς άλλους είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, δανείων των Ιρλανδικών τραπεζών ω το Σεπτέμβριο του 2008 και όλα αυτά τα οποία είχαμε στα χέρια μα τότε δεν καταδεικνύαν το μέγεθο του προβλήματο. Γιατί όλα, όλη η καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού αφορούσαν τι ε, τιμές των ακινήτων, οι οποίε πριν από έξι μήνε ήταν ακόμα υγιείς. Δεν ήταν λοιπόν εκτός αν ήταν κανείς προφήτης να φανταστεί, να φανταστεί ότι θα υπήρχε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και φανταζόταν θα υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Καταλαβαίνω που λέτε για την κρίση, για την κατάρρευση της Lehman Brothers, ότι ήταν μια προβλέψιμη κρίση. Αλλά αν ήταν τόσο προβλέψιμη, γιατί έγινε τόσο γρήγορη η κατάρρευση σε τόσα μέρη συγχρόνως και μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ήταν τόσο εύκολο να την προβλέψει κανείς τότε όσο είναι τώρα εκ των υστέρων να τα δει κανείς. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους κεντρικούς τραπεζίτες για το ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συνέβαινε τότε. Το 2008 δεν είχαμε λοιπόν υπόψη μας όλους τους κινδύνους για την οικονομία. Δεν περιμέναμε ότι και οι έξι κύριοι κίνδυνοι για την οικονομία θα εμφανιζόντουσαν συγχρόνω Από την εμπειρία μου στο χρηματοπιστωτικό τομέα πριν από την κρίση, νομίζω ότι οι εκθέσεις έδειχναν ότι το Υπουργείο Οικονομικών έδινε σαφή μηνύματα για τον κίνδυνο της υπερθέρμανσης της οικονομίας. Κάθε φορά που λέγαμε βέβαια ότι υπήρχε κίνδυνος υπερθέρμανσης της οικονομίας, τον επόμενο χρόνο μας διέψευδε η οικονομία, που είναι πολύ καλύτερα από τον προηγούμενο χρόνο. Επομένως δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους υπουργού που δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ανάγκη προσαρμογής οικονομίας. Οι περισσότερες προβλέψεις έλεγαν ότι εν καιρό θα χρειαστεί προσαρμογή, αλλά όχι του χρόνου. Για το ερώτημα της κυρίας Childers, γιατί με, με διορίσαν στη θέση αυτή, συγγνώμη που περί αυτολογώ σε αυτή την περίπτωση, αλλά η κυβέρνηση με έθεσε σε αυτή τη θέση, διότι πιστεύω ότι ήθελα να εξασφαλίσουμε ότι θα είχε σωστή εκπροσώπηση η Ιρλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμβολή της Ιρλανδίας συμπεριλαμβάνει και το διορισμό των σωστών ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τι περνάει από το κεφάλι του, των Υπουργών και των κυβερνητών κάθε χώρας αλλά εγώ θεώρησα ότι ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα το ότι με διορίσανε. Και μετά από τις εικασίες που δημιουργήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης, σκέφτηκα και εγώ ότι ίσως αυτό να γίνει πιθανό. Μου λέτε τώρα πώς περιέγραψα αυτή την εργασία, σύμφωνα με τις εφημερίδες. Αυτό το οποίο δεν είπαν οι εφημερίδες είναι ότι μετά από τέσσερις, τέσσερα έτη αγώνα που κάνει κανείς κάθε μέρα τη σκέψη μήπω έχω κάνει ένα λάθος που θα στοιχήσει σε ένα δισεκατομμύριο. Σε σχέση με αυτό το Ηράκλειο σχεδόν έργο, θεώρησα ότι αυτό που έχω να κάνω τώρα στο ελεκτικό συνέδριο θα είναι πανεύκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πεδαριώδε το έργο του ελεκτικού συνέδριου. Okay, we go to the next. Επόμενος γύρος, ζεύγους δύο, τριών ερωτήσεων. Κύριος Κλάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ήθελα να ζητήσω εκ μέρου συνδέλφων που δεν είναι σήμερα παρόντε, συγγνώμη. Κύριε Κάρντιφ, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Οικονομικών, ήσασταν υπεύθυνο για ένα σοβαρό σφάλμα 3,6 δι. Ήταν 1,8 τα δισεκατομμύρια ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς ήταν το πρόβλημα και η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο το διπλασίασε και άφησε να πιστέψουμε πως αυτό ήταν το χρέος. Όταν ήσασταν υπάλληλο δε, ε, εσείς δώσατε συμβουλή στην κυβέρνηση να οδηγήσει, ε, να επιτρέψει την ε, πτώχευση τραπεζών οι οποίες άφησαν εκατομμύρια ανθρώπους ε, ε, χωρίς φράγκο. Με... Γιατί δεν το κάνατε αυτό, ενώ οι συμπολίτες σας έπρεπε να υποφέρουν από λιτότητα, δυσκολίες και αυτό για χρήματα τα οποία εσείς χειριστήκατε λάθος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντερόσα που με ενημέρωσε και που έθεσε ερώτηση για την οποία εγώ δεν ήμουν ανήμορος. Να έρθω στο θέμα της ευθύνης και της λογοδοσίας. Ο κύριος Κάρδιφ απαντά στις ερωτήσεις που του τίθενται στην, ε, στην συνέντευξη αυτή. Όταν ε, μίλησε για τα χαρακτηριστικά της υγιούς ε, διακυβέρνησης και του δημόσιου τομέα, ε, είπε ότι η λογοδοσία είναι θέμα κλειδί. Σε σχέση με το 3,6 δις, θεωρεί δηλαδή ότι η λογοδοσία για τα σφάλματα που έγιναν μεταφέρεται μέχρι και στους διευθυντές οι οποίοι ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι εκείνοι. ή μήπως αυτόματα βαραίνουν τον Γενικό Γραμματέα. Και ιδιαίτερα καθώς ο Γενικός Γραμματέας κάθε Υπουργείο στην Ιρλανδία έπαιρνε αμοιβέ πάνω από αυτές του Πρωθυπουργού. Πώς λοιπόν το συνδυάζει αυτό με το ότι δεν δέχεται την ευθύνη στο επίπεδο του Γενικού Γραμματέα για τα σφάλματα που έγιναν και τα μεταφέρει τα σφάλματα αυτά στους ώμους των διαφόρων διοικητικών επιπέδων. Εφόσον λοιπόν έγινε ευεσφάλμα, ποιος είναι αυτός που είναι υπεύθυνο, ιδιαίτερα εν ώψη της απάντησης που μας έδωσες στις ε, ερωτήσεις αυτές που του έγιναν. Διαφάνεια και λογοδασία των διευθυντών είναι θέμα κλειδί. Είναι πολύ βασική. Σας ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Οντί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση κύριε Πρόεδρε γιατί Έχουμε εδώ μια ολόκληρη σειρά ερωταπαντήσεων και δεν είμαι βέβαιος πως τα έγγραφα που έχουμε συν αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα αρκέσουν για μας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε πλήρη γνώση του θέματος. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κάρδιφ. Η συνθήκη προβλέπει ότι τα μέλη της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου θα είτε θα πρέπει να έχουν συμμετέχει στο θεσμό εξωτερικού ελέγχου του κράτους τους ή να έχουν ιδιαίτερα προσόντα στον, ε, όσον αφορά τον έλεγχο. Εσείς διατελέσατε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών με πολύ υπεύθυνε θέσεις ε, στο, και αρμοδιότητες, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προσόντα σας όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο. Ποια είναι η φύση των προσόντων σας λοιπόν που θα μας επέτρεπε να έχουμε θετική γνώμη για το άτομό σας. Και έπειτα, όταν συγκρίνω το σύνολο των mail που λάβαμε σε σχέση με το ερωτηματολόγιο, γιατί υπήρξε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απέφυγε η γραμματεία μας στον υποψήφιο για κλασικά ερωτήματα. Αυτές οι ερωτήσεις συν αυτήν την ακρόαση θεωρώ πως δεν είναι επαρκής. Και τώρα κάνω ένα διαδικαστικό θέμα, τη παρουσία του υποψηφίου, μήπως θα έπρεπε μετά από αυτές τις ερωτήσεις, συν τις ερωτήσεις που λάβαμε από τους πολίτες, συμπολίτες μας, γιατί αυτούς αντιπροσωπεύουμε εδώ, να υπάρξει ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο κάπως πιο τεχνικής φύσης, ίσως και πιο πολιτικής φύσης, το οποίο θα απαντούσατε γραπτός για να δούμε ακριβώς ε, που βρισκόμαστε και να συνοψίσω τη θέση μου εφόσον υπήρξαν σφάλματα Εντάξει, εγώ συχνά λέω και στα παιδιά μου πως η εμπειρία είναι το σύνολο των λαθών. Δεν έγιναν μόνο στην Ιρλανδία λάθη, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Πάντως αυτό που δεν δέχομαι είναι να μας ε, οδηγήσουν σε σφάλμα. Δεν θα έλεγα ότι ψεύδεται κανείς, αλλά εμείς χρειάζεται να γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Πέρασαν από εδώ υποψήφοι άλλων χωρών που είχαμε την αίσθηση ότι δεν μας έλεγαν την αλήθεια, είχαμε δύσκολες ψηφοφορίες στην Ολομέλεια και θα ήθελα πολύ να γίνει μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων και να μπορέσετε να μας απαντήσετε συγκεκριμένα και γραπτό σε όλα τα τεχνικά ερωτήματα που μας έθεσαν οι πολίτες για να γνωρίζουμε τελικά στην ουσία ποιο είστε, γιατί εγώ δυσκολεύομαι να σχηματίσω άποψη. Πρόεδρε, και ήθελα αυτό να το πω. Κύριε Κάρντιφ, μπορείτε να προσπαθήσετε να απαντήσετε μέσα σε τρία λεπτά. Um, Θα κάνω ό,τι μπορώ, Πρόεδρε. Uh, on the misstatement, um issue, uh, um, I think Κύριε Κλάρκ, νομίζω πως το απάντησα αυτό που είπατε. Εγώ είπατε, συμβούλεψα την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι είπα στην κυβέρνηση, αλλά έδωσα στην κυβέρνηση μια σειρά επιλογών. Δεν υπήρχε καμία συγκεκριμένη εγγύηση, παρά μόνο μια πολύ ευρεία εγγύηση οι επιλογές που έδωσε στην κυβέρνηση συμπεριλάμβαναν και μια ολόκληρη σειρά άλλων επιλογών και δόθηκαν στους αρμόδιους υπουργούς οι συμβουλές αυτές και ειλικρινά δεν δέχομαι ότι οδήγησα τον Ιρλανδικό λαό στην πτώχευση και σίγουρα δεν ήμουν ο μόνος άνθρωπος που έδωσα συμβουλές περί αυτού στην κυβέρνηση. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Κέλλη για το ότι δεν βαραίνει, ότι μάλλον η ευθύνη βαραίνει το Γενικό Γραμματέα και ότι δεν βαραίνει τους όμως των υπολείπων ε, υφιστάμενων, δεν πάει πάντα έτσι κύριε Κέλλη. Είμαστε της γενικής άποψης και μάλιστα και εδώ προσπάθησα να αποφύγω τον ε, μπω σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά θα μπορούσε να συμβεί λόγω της πίεσης υπό την οποία εργαζόμαστε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος να κάνει λάθος ε, υπό συγκεκριμένη πίεση, υπό ε, πίεση και ανθρωπίνων ε, πόρων. Οι μισθοί υπήρξαν ψηλοί στην Ιρλανδία. Μπορεί να ήταν ψηλότερη μισθή από του Πρωθυπουργού, είπατε, αλλά δεν ήταν δύο φορές ο Πρωθυπουργός μείωσε τον μισθό του και α, ταυτόχρονα το έκανα και εγώ. Οπότε ποτέ δεν πήρα περισσότερο μισθό από τον Πρωθυπουργό. Τώρα, εγώ προσπάθησα να μην κατηγορήσω άλλος ειλικρινά, παρά ανοιχτά να συζητήσω με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές κάθε φορά πολύ σύντομα μετά από τα, γεγονότα ώστε να εξηγήσω όσο γινόταν καλύτερα τα συμβάντα όσον αφορά τα περαιτέρω ερωτηματολόγια και ούτω καθεξής εσείς ε, και το είπατε αυτό κύριε Οντία αλλά αυτό είναι θέμα της Επιτροπής σας όχι δικό μου ο διερμηνέας χρησιμοποίησε τη λέξη αλήθεια και μπορώ να σας πω ειλικρινά πως προσπαθώ να σας πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Thank you. Congratulations. Πολύ ωραία. Τρία λεπτά ακριβώ. Οι τελευταίοι ομιλητές είναι καταρχήν ο κύριος Ντερόσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κύριε Κάρντιφ στην σημερινή μας ακρόαση θα ήθελα να πω εκ προημίου που χαίρομαι πάρα πολύ που η Ιρλανδική κυβέρνηση προσφέρει σε ένα άτομο τέτοιου επίπεδου, τέτοιου, τέτοιων προσόντων και τέτοια ακαιρεότητα στη θέση αυτή στο ελεκτικό συνέδριο. Για πολλές φορές εγώ συζητούσα με τους συναδέλφους μου στην κυβέρνηση και τόνισα ότι πρέπει να κάνουμε ε, μια πραγματική συμβολή στην Ευρώπη και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μονάχα στέλνοντα τα άτομα που έχουν τα υψηλότερα δυνατά προσόντα. Και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον με ακούσαν και προτείναν τον κύριο Κάρδιφ για αυτή τη θέση. Με εντυπωσιάζει ο ανοιχτό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα ερωτήματα που σα τίθενται, κύριε Κάρδιφ. Και θα ήθελα να παροτρύνω τα μέλη της Επιτροπής μας να μην δίνουν σημασία σε email τα οποία κινούνται από ε, πολιτικές ιστεροβουλίες και να κοιτάξουν μονάχα τα πραγματικά γεγονότα, τα προσόντα και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που έλκουμε από τις συνθήκες, να, να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που διορίζουμε έχουν τα προσόντα, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία που απαιτούνται. <clears throat> Θα ήθελα να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα στον κύριο Κάρτιφ για την έκθεση Χόνεμπορ νομίζω ότι γνωρίζετε, είναι μια έκθεση που έχει να κάνει με την τραπεζική κρίση. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε ότι η έκθεση Χόνεβο έκανε σαφές ότι η κρίση στην Ιρλανδία ήταν απόρρια συστημικών προβλημάτων και τα προβλήματα αυτά είχαν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο δεν λειτουργήσε σωστά η ρυθμιστική λειτουργία, ότι οι ρυθμιστικές αρχές της Κεντρικής Τράπεζας και των χρηματοπιστωτικών τομέων δεν χρησιμοποιηθήκαν πλήρως οι εξουσίες αυτές και προέκυψαν προβλήματα αυτού του είδους σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες λόγω μιας συγκεκριμένης προσέγγισης προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Κάρντιφ. Εγώ έρχομαι με ανοιχτό μυαλό σε αυτή την ακρόαση και θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο κ. Ντερόσα. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά ανοιχτέ και τίμιε οι ειλικρινεί οι απαντήσει σα. Δεν <clears throat> κάνετε τον πόντιο και τον πιλάτο ύπτοντα στα χέρια σα, ούτε προσπαθείτε να προστατεύσετε την κυβέρνησή σα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιε αποφάσει οι οποίε έχουν να κάνουν με πολλού φορεί και την Κεντρική Τράπεζα και εξωτερικέ δυνάμει. Δεν ήταν εύκολο λοιπόν να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι μακρά η ιστορία της κρίσης. Τα ερωτήματά μου τώρα, στην απάντησή σας στο ερώτημα 10, είπατε ότι η έλεγχοι απόδοσης δίνει τη δυνατότητα στους φορείς να έχουν καλύτερες πληροφορίες από αυτούς τους ελέγχους επίδοσης. Ποια είναι λοιπόν η εμπειρία που αποκτήσατε, αποκομίσατε κατά τη διάρκεια τη κρίση τη Ιρλανδία. Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα στη θητεία σα στο ελεκτικό συνέδριο. Δεύτερον, ο πρωταρχικό ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου να εξετάζει κατά πόσον έχει εφαρμοστεί σωστά ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουν χρησιμοποιηθεί με σωστή διαχείριση τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τι ανησυχίε που ακούσαμε σήμερα και δεν θα πω τώρα στι λεπτομέρειε, πώ θα απαντούσατε για το κατά πόσο η δική σας κυβέρνηση πράγματι έκανε σωστή διαχείριση στη χειρότερη εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τέλος κύριε Κάρδιφ, το πρώτο ερώτημα που θα σας έθετα αν θα σας πρόσφερα εγώ μια εργασία, μια θέση εργασίας, θα σας ρωτήσω γιατί θεωρείτε ότι είστε καλός υποψήφιος για το ελεκτικό συνέδριο. Κύριος Γκέλαχερ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπα, <clears throat> θέλω να πω μάλλον καταρχήν, ότι παρά την ε, δημοσιότητα που περιτριγυρίζει την ε, υποψηφιότητα του κυρίου Κάρντιφ, εγώ έρχομαι εδώ πέρα με ανοιχτό πνεύμα σε σχέση με αυτό το θέμα. Το ερώτημα μου τώρα, πώς θα μπορούσε η συνεργασία μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου, των Εθνικών Ελεκτικών Φορέων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ελέγχου του προπολογισμού, πώ θα μπορούσε να βελτιωθεί κατά την άποψή σα και πώ θα βλέπατε τα καθήκοντά σα για την. Ε, για το να δίνετε εκθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά τα δημοσιονομικά. Ε, εσείς είσαστε υποχρεωμένοι από τη συνθήκη να βοηθήσετε το, ελεκτικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει εξουσίες του σε σχέση με τον έλεγχο των δαπανών. Δύο τελευταία στιγμή είπαν ότι θέλουν να μιλήσουν. Είχα κλείσει τον κατάλογο, αλλά θα ήθελα όλοι να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Η κυρία Γκρέσλερ και η κυρία Μαγκίνες να θέσουν ένα ερώτημα, αλλά ενός λεπτού και μόνο. Ingeborg. Ich möchte auf ein... Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 για τις συνέπειες της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης σε ό,τι αφορά το δημόσιο έλεγχο των δημοσιονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου, όπου και αναφέρεται ότι δεν έχει αρμοδιότητε ε, το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά θα ήθελε να έχει αρμοδιότητε σε ό,τι αφορά την, ε, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διάσωση. Συμφωνούμε με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο απόλυτα. Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο δημοσιονομικό έλεγχο θα πρέπει να υπάρχει από πλευρά του λεκτικού συνεδρίου. Ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει σύγκρουση ε, σε ό,τι αφορά το ρόλο σα στο λεκτικό συνέδριο και στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ και τέλο, η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ πρόεδρε που δείχνετε και κατανόηση γιατί καθυστέρησα στην ακρόαση. ορίζω τον κύριο Κάρντιφ από πλευρά τη γεωργική πολιτική. Έχω να το εξή από πρακτική άποψη γιατί τέθησα, ακούσαμε και πολιτικές ερωτήσεις. Όταν μιλάμε στους αγρότες, στην επικράτητά μας, υπάρχει ο φόβος ε, του ελεγκτή. Θεωρώ ότι χρειάζεται έλεγχος των δημοσιονομικών δαπανών, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τα δικά σας σχόλια σε ό,τι αφορά μια πολιτική γεωργικής ε, φύσεως. Μήπως θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε στους ελέγχους να καταστούν αρκετά ευέλικτοι ε, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις μεμονωμένες συνθήκες πληρώντα ωστόσο τα κριτήρια που έχουμε θέσει στο Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί φοβάμαι ότι με τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ θα καταλήξουμε να είμαστε πιο παγιδευμένοι. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να καταλάβει κάποιε από τι ε, συνέπειε του έργου αυτού. Ευχαριστώ. Κύριε Κάρτιφ, έχετε το λόγο. Σας δίνω τέσσερα λεπτά αυτή τη φορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Ντερόσα για τα σχόλιά του, τα οποία τα εκτιμώ ιδιαίτερα. Η ερώτησή του για την έκθεση χώμα. Νομίζω ότι σωστά την ερμήνευσε. Ξέρετε ότι πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο και ασφαλώς αν γίνονται κάποια λάθη θα πρέπει να τα εξετάζουν τελικά τα υπουργεία και στην Ευρώπη πάντα επιμένουμε τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες να είναι πιο ανεξάρτητοι οι νομοθέτες, αλλά τελικά δεν ελέγχουμε κατά πόσο κάνουν τη δουλειά τους σε δεύτερο βήμα. Στην ε, Ιρλανδία η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, εκτός από το τομείς που δεν υπήρχε κρίση, ε, εκτιμήθηκε από το IMF από το είμαι Νομισματικό Ταμείο. Πώς θα εξετάσουμε λοιπόν το έργο των νομοθετών, με ποια κριτήρια θεωρούσαν ότι ήταν καλό το έργο του τότε, ότι ήταν καλές οι εκθέσεις, αλλά με την πρόσφατη νομοθεσία καταλάβαμε ότι είχαμε εφαρμόσει μία ε, νομοθεσία και ότι η... καταλάβαμε ότι οι Ευρωπαϊκοί ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να ελέγχονται και να ελέγχουν το έργο των νομοθετών. Για το ερώτημα της κυρίας Χάρκιν για την καλή διαχείριση και το καθεξής και κατά πόσο είμαι καλό υποψήφιο. Είμαι καλό υποψήφιο, όχι μόνο επειδή διαχειρίστηκα μία κρίση, αλλά είναι ανοιχτή και ειλικρινή η προσέγγιση μου στη δουλειά. Έχω κυριότητα σε όλη μου τη δουλειά. Δεν ασκώ πίεση, ακόμα και όταν λαμβάνω χιλιάδες email. Δεν κάνω πίσω και ασφαλώς δεν ψεύδομαι. Άρα έχω θεωρώ μεγάλη προσωπική ακεραιότητα και δεύτερον έχω σημαντική εμπειρία στη διοίκηση τουλάχιστον ενός οργανισμού, όχι μόνο σε περίοδους κρίσης, γιατί ήμουν υπεύθυνο ε, για το διοικητικό προϋπολογισμό της ε, υπηρεσίας ε, δημοσίων υπαλλέλων. Έχω καλή εκτίμηση των ε, περιορισμών και των δυνατοτήτων των ε, δημοσίων υπηρεσιών και ξέρω που μπορεί να ανακύψουν ζητήματα. Για το πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με εντυπωσίασε την τελευταία εβδομάδα η ετήσια έκθεση. Ήταν καλό παράδειγμα όπου το Συμβούλιο και το Συνέδριο μαζί με την Επιτροπή η Επιτροπή επεσήμανε τομείς όπου καταβάλλονταν πραγματικές προσπάθειες για να βελτιωθεί η λειτουργία της σε ό,τι αφορά ε, τον έλεγχο και σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα του Κοινοβουλίου ως προς τον έλεγχο. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι καλό παράδειγμα. Είναι σαφές ότι το 2005 υπήρξε μία έκθεση και έγιναν πολλές συστάσεις βάσει των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι προς το κοινό μας ε, συμφέρον, αλλά το πλεονέκτημα του Κοινοβουλίου και εδώ επανερχόμαστε σε θέματα αξιολόγησης σε τακτικά διαστήματα, οι στόχοι ενός προγράμματος δεν είχαν ε, διευκρινιστεί αρκετά σαφώς προκειμένου να ε, έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εμείς ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, είτε ως πολιτικοί είτε ως σύμβουλοι, θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς τους στόχους, προκειμένου να επιτρέψουμε τη διεξαγωγή σωστών ελέγχων και σωστού σωστής αξιολόγησης. Άρα πιστεύω ειλικρινά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάδραση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και σε επίσημο και σε ανεπίσημο επίπεδο. Το βασικό και το κρίσιμο στοιχείο φυσικά είναι να θέσουμε προτεραιότητε για το τι θα πρέπει να περνάει από έλεγχο. Γιατί φυσικά υπάρχει τεράστιο όγκο σε ό,τι αφορά την ε, ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση υπάρχει μια θεσμική κρίση ασφαλώς και ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό το κοινό να εκπροσωπείται σωστά στον έλεγχο στο πλαίσιο των θεσμικών ε, οργάνων. Το θεσμικό πλαίσιο μάλλον δεν ε, επιτρέπει στο ελεκτικό συνέδριο να αναμειχνύεται στα, σε όλα τα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι θα προβλεφθούν περαιτέρω αρμόδια για την κυρία Μαγκίνες τώρα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την κατάσταση των αγροτών. Θεωρώ ότι ο αγρότης του οποίου η Ελλάδα επιλέχθηκε δειγματοληπτικά, επειδή υπάρχει και ο γεωργικός ελεγκτής, πιστεύω ότι το βασικό και εδώ είναι σαφής στόχη ως προς την πολιτική και σαφείς προδιαγραφές για το κάθε άτομο. Γιατί αν δεν είναι σαφείς και ξεκάθαροι οι κανόνες, πώς είναι δυνατόν ο κόσμος που δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοια χαρτούρα να καταλάβει τι χρειάζεται. Χρειάζεται λοιπόν σαφήνεια για καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η ακρόαση, αλλά θα πρέπει φυσικά να πάρει το λόγο και η εισηγήτρια για να συνοψίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια κλείνοντα. Να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τι παρατηρήσει του και για τι ερωτήσει που έθεσαν. Θα προσπαθήσω να σα βοηθήσω να λάβετε μια απόφαση σε τέτοιε ακροάσει. Ένα από του συναδέλφου έκανε σχετικέ προτάσει έχουμε κι άλλα στοιχεία αξιολόγησης σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους, τους οποίους εξετάσαμε σήμερα το πρωί, όπου ορισμένοι δεν έθεσαν αυτή την διάσταση του, της ακρόασης. Ε, στην περίπτωση του κυρίου Κάρτιφ και στην περίπτωση του Ιρλανδικού συστήματος, ο ελέγχος των τραπεζών ε, έγινε από μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Αυτό ισχύει και για την Κεντρική τράπεζα που ήταν και αυτή ανεξάρτητη. Άρα ο κύριος Κάρντιφ δεν μπορούσε να διεξάγει παράλληλα έλεγχο και να συμμετάσχει να συμμετέχει και στις ε, διαβουλεύσεις της ε, κυβέρνησης. Ε. Έχουμε τον κύριο Μαγκρίβη, ο οποίος δεν είχε κάποιο ενδιαφέρον να ρυθμίσει την τραπεζική κρίση. ζητήθηκε από την ανάλογη Ιρλανδική Ιεραρχία να λάβει τις σχετικές αποφάσεις και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι πρόκειται σε κάθε περίπτωση για ένα συστημικό λάθος, το οποίο δεν έχει να κάνει με προσωπική ευθύνη αυτό. Δεν το λέω μόνο στον κύριο Κάρτεφ, το λέω και σε άλλους. Το λέω και για τους αρμόδιους πολιτικούς, τους αρμόδιους υπουργούς, εκείνους οι οποίοι είχαν εκλεχθεί Όπω σημαίνει συχνά με τέτοιε πολιτικές αποφάσεις. Κάτι επιπλέον θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσω από τους συναδέλφους να επιτύξουν προσοχή. Δεν ξέρω πόσα email λάβατε, ίσως κάποιες χιλιάδες, ίσως και κάποιες δεκάδες. Δεν θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να πέσει η σκιά, αν θέλετε, ενό άλλου μέλου του ελεγκτικού συνεδρίου πάνω σε αυτόν τον υποψήφιο. Αυτό θεωρώ ότι δεν θα ήταν. Ε, δεν είναι, είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να δούμε και να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτή η πολιτική εκστρατεία είχε να κάνει με τον ε, υποψήφιο. Εδώ ερωτούμε ένα συγκεκριμένο υποψήφιο για το κατά πόσο ε, διατίθεται για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει προταθεί. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να είμαστε ψυχροί αν θέλετε και αμερόληπτοι σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των email που λάβαμε γιατί αποτελούν και αντιδράσεις στην τραπεζική, τραπεζική κρίση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προσωπική ευθύνη, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν συστημικά προβλήματα σε ό,τι αφορά το μηχανισμό διάσωσης, ο οποίος ισχύει ισχύ, Και πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται προσπάθειες να εξέλθουμε τις κρίσεις αυτής. Υπάρχουν άτομα τα οποία φυσικά ε, ε, δεν ευθύνονταν για την κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάρντιφ και διακόπτω για λίγα λεπτά την συνεδρίαση προκειμένου να προσέλθει ο υποψήφιος από την Ιταλία. May I ask everybody to... Σας παρακαλώ καθίστε πάλι γιατί θα συνεχίσουμε. Όσοι θέλουν να συζητήσουν να σπάνε στο καφενείο. may I once again ask you to have your conversations in another place than here? Then I open this. Ξεκινάμε την συνεδρίαση και πάλι. Να καλωσορίσω τον κύριο Πιέτρο Ρούσο που έχει οριστεί από την Ιταλική κυβέρνηση The court of... και υποψήφιος για το ελεγκτικό συνέδριο. Όπως ο κύριος ε, Ρούσο θα έχει το λόγο για πέντε λεπτά περίπου, όπως και οι άλλοι υποψήφοι, για να μας εξηγήσει γιατί θέλει να γίνει μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου και τι σκοπεύει να κάνει και έχετε το λόγο κύριε ε, Ρούσο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας ως Ιταλός υποψήφιος για τη θέση του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε αυτή μου την παρέμβαση δεν θα σας μιλήσω για σταδιοδρομία μου, την οποία ήδη γνωρίζετε μέσω του βιογραφικού σημειώματος που σας έχω υποβάλει. Παρά μόνο να πω και να υπογραμμίσω ότι η επαγγελματική μου πορεία αποτελείται από την υπηρεσία που έχω προσφέρει ως εισαγγελέα και για τη μεγαλύτερη διάρκεια της υπηρεσίας μου ως εισαγγελέα του Ιταλικού Ελεκτικού Συνεδρίου, δηλαδή στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου της δημόσιας οικονομίας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη θέση μου σε σχέση με την άσκηση της, ε, του λειτουργήματος του μέλους του Ελληνικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους λόγους για τους οποίους είμαι πεπισμένος ότι μπορώ να προσθέσω κάτι ε, με τα δικά μου προσόντα στις δραστηριότητε αυτού του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου. Φυσικά είμαι έτοιμος να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση που θα μου θέσετε σε σχέση με τις δραστηριότητες που έχω ε, ασκήσει μέχρι τώρα. Η άσκηση αυτής της ε, πολύ σημαντικής θέσης θα αποτελέσει το αποκορύφωμα για την σταδιοδρομία μου. Η λειτουργία του εισαγγελέα που είχα μέχρι τώρα ε, συνίσταται στην εφαρμογή της νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη δραστηριότητα των ε, δικαστών λογιστών στην επαγρύπνηση για τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος από πλευράς του διοικητικού μηχανισμού που στηρίζει τις δράσεις ε, του πολιτικού οργάνου που άμεσα εκλέγεται από τους πολίτες. Γνωρίζω λοιπόν πάρα πολύ καλά τις ευθύνες που βαραίνουν ε, τους ε, συμμετέχοντες στο θεσμικό αυτό όργανο που δικαίως έχει οριστεί ως ε, η δημοσιονομική συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ασκεί το ρόλο αυτό μέσω της ελεκτικής του δραστηριότητα όσο και δίνοντας το παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα. Όσον αφορά, μάλλον καθώς έχει αναλάβει την προστασία των χρημάτων των πολιτών, το όργανο αυτό αποτελεί το ύπατο ε, όργανο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θεωρώ ότι χάρη στην προσωπική μου εμπειρία στο ε, ελεγκτικό συνέδριο και στον έλεγχο της δημόσιας οικονομίας της χώρας μου, Πιστεύω πως μπορώ να συμβάλλω θετικά στις δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον και την προστασία των ε, οικονομικών της Ένωσης. Ε, φυσικά ξέρω ότι είναι πολλές οι δεσμεύσεις και οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσω σε μια τόσο ευαίσθητη συγκυρία όπως η σημερινή απέναντι στην παγκόσμια κρίση που, έχει, που μαστίζει τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και που ε, επίσης πλήττει τις δημόσιες οικονομίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ε, προσεκτική στην κινητοποίηση και τη χρήση των πόρων της για λογαριασμό των πολιτών και των φορολογουμένων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το έργο του εξωτερικού ελεγκτή της δημόσιας οικονομίας σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικός και κρίσιμος και αποκτά κρίσιμη ε, ακόμα μεγαλύτερη σημασία μέσα στον ε, θεσμικό μηχανισμό. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των αρμοδιοτήτων είναι, όπως είπα, το να λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τις νομοθετικές, ε, τα νομοθετικά σώματα που αντιπροσωπεύουν άμεσα τον λαό και την κυριαρχία του και στα οποία σώματα, στα δημοκρατικά καθεστώτα, ε, ανήκει η τελική αξιολόγηση της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ο σύνδεσμος αυτός είναι ιδιαίτερα προφανής από τις ίδιες υποθέσεις που οδήγησαν στην γέννηση αυτού του σώματος. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που η, το θεσμικό όργανο του Ελληνικού Συνεδρίου μέσω της, ε, της συνθήκης των Βρυξελών του 1975 κατέστη μάλλον η δημιουργία του συνεδρίου έγινε ταυτόχρονα με την εισήγηση των ιδίων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την απόδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου σημαντικών αρμοδιοτήτων σε θέματα προπολογισμού. Θα ήθελα να θυμίσω ότι ο Χάρι Χάγνερ, που ήταν στο παρελθόν Πρόεδρο τη Κομισιόν για τον έλεγχο του προπολογισμού, από τι αρχέ του 1970 αγωνίστηκε για τη δημιουργία ενό ελεγκτικού ανεξάρτητου οργάνου ε, για την κοινοτική οικονομία όπου αυτό αποτελεί ένα διάστο σύμβολο της ανάγκης ε, για σχέση συνεργασίας ανάμεσα στο Ελληνικό Συνέδριο και το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με αυτήν εδώ την Επιτροπή συνεργασία που ήταν ε, πολύ, πολύ αποτελεσματική και που μπορεί περαιτέρω να ενισχυθεί. Για μένα είναι κίνητρο η σκέψη του να μπορώ να συμμετέχω στις δραστηριότητες μιας, ε, ενός θεσμικού οργάνου που έχει τόσο σημαντικό έργο, δίνοντας τη δική μου συμβολή στην συγχώνευση αυτή των διαφόρων πολιτισμών που βρίσκεται στην βάση του ίδιου του πνεύματος της Ένωσης και αποτελεί και την ισχύ της. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι στηριγμένο στη δική σας εμπιστοσύνη θα τελέσω τα καθήκοντά μου με απόλυτη ανεξαρτησία, ακαιρεότητα και διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρούσο και τώρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για να κάνει τη δική της ε, εισήγηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Ρούσο, καλώς ήρθατε κύριε Ρούσο. Επιτρέψτε μου να σας θέσω κάποια ερωτήματα που μπορεί να σας εκπλήξουν, αλλά που έχουν να κάνουν με τις συζητήσεις που κάναμε σήμερα εδώ πέρα. Προταθείτε, πρώτα προταθήκατε ως υποψήφιος από την, από την Ιταλική κυβέρνηση. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση, η κυβέρνηση που σας πρότεινε του κυρίου Μπερλουσκόνη ή του κυρίου Μόντι. Δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω, στην τελευταία απάντηση που δίνετε στο τελευταίο ερώτημα, όταν σας ρωτάμε αν το Κοινοβούλιο έλεγε ότι δεν σας εγκρίνει, δεν είναι σαφές από τη δική σας απάντηση, ίσως είναι θέμα μετάφρασης, δεν είναι φανερό αν εσείς θα αποφασίζετε να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας. Γιατί λέτε ότι θα ρωτούσατε την Ιταλική κυβέρνηση, που θα είναι πια η κυβέρνηση του κυρίου Μόντσι, που δεν νομίζω ότι είναι αυτή που σας προέτεινε. Ε, ένα άλλο θέμα πιο πολύ ουσίας. Έχετε ένα ενδιαφέρον προφίλ για το ελεκτικό συνέδριο και ήσασταν ήδη μέρος του Ιταλικού Ελεκτικού Συνεδρίου και έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την άμυνα που είναι ένας σημαντικός τομέας και ιδίω με τα θέματα δημοσίων προμηθειών και ήθελα να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Έχετε συμμετάσχει σε μία και αναφέρεται σε μια σημαντική στιγμή της καριέρας σας το γεγονός ότι συμμετάσχατε σε ένα έλεγχο του Ιταλικού Υπουργείου Άμυνας όπου είχε υπάρξει ένα πρόβλημα για την ε, ενοικίαση αμερικανικών αεροσκαφών πριν από το Eurofighter και είπατε ότι αφορούσε σημαντικά κονδύλια. Είπατε ότι συμμετάσχατε στην απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό όμως δεν καταλαβαίνω είναι αν οι αποφάσεις σας οδήγησαν σε μία εξοικονόμηση, βελτίωση των δημοσίων προμηθειών ή οτιδήποτε άλλο. Ένα από τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίσουμε και τώρα γίνεται πιο ανάγλυφο, το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν όλο και περισσότερη ευθύνη και συμμετέχουν με σωστό τρόπο στον στην συνεργασία των προϋπολογισμών θα πρόκειται για προϋπολογισμούς όπου συμμετέχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια. Πώς θα μπορούσατε λοιπόν από ένα ευρωπαϊκό ελεκτικό συνέδριο να βελτιώσετε αυτή τη συνεργασία με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια για να αναδυθεί μια δυναμική μέσω της οποίας το Συμβούλιο των Υπουργών θα μπορούσε να βελτιώσει την υπευθυνοποίησή του έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αν μπορείτε να απαντήσετε στα αγγλικά ή στα γαλλικά κάποια από αυτέ τι δύο γλωσσε που νομίζω ότι γνωρίζετε εξαίρετα. <laughs> Θα απαντήσω σε, ένα άλλο, σε μια άλλη γλώσσα, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να σα ευχαριστήσω για το ερώτημά σα και μιλάτε και μιλήσατε για πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα. Θα Συνεχίζω στα γαλλικά τώρα. Η πρώτη ερώτηση που θέσατε αφορά την, τον διορισμό μου από μια κυβέρνηση η οποία πια δεν είναι, δεν είναι πια στην εξουσία. Έχουμε μια κατάσταση ιδιαίτερη στην Ιρλανδία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διορισμού των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Δεν υπάρχουν έγγραφες, προδιαγραφές για κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια εθνική διαδικασία η οποία έχει ακολουθηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και η οποία κατά την απόψή μου εξασφαλίζει το μη πολιτικό χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας. Μετά από το διορισμό του πρώτου μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση έχει περιοριστεί να ζητά από το Ιταλικό Ελεκτικό Συνέδριο να καθορίζει ένα δικαστικό για την θέση αυτή και πάντα το Ιταλικό Ελεκτικό Συνέδριο έχει θέσει μια τέτοια προτείνη όχι τόσο μέσω της απόφασης του Προέδρου του, αλλά με ένα εσωτερικό διαγωνισμό, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά κανόνων και μπορώ να σας δώσω όλες τις ε, τυπικές υποχρεώσεις των υποψηφίων στη δική μου περίπτωση και πάντα γίνεται λοιπόν μια πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος ε, μέσα στα πλαίσια του ελεκτικού συνεδρίου μεταξύ όλων των δικαστικών και πάντα υπήρχε αυτή η επιλογή του υποψηφίου βάσει τίτλων και σε σχέση με κριτήρια τα οποία είχαν εκ των προτέρων καθοριστεί. παραδείγματος χάρη το θέμα της ε, αρχαιότητος στην καριέρα του. Με ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με την καριέρα αυτή και τις υπευθυνότητες που έχει αντιμετωπίσει ο καθένας. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και στη δική μου, η Ιταλική κυβέρνηση πάντα λάμβανε την υποψηφιότητα από το ελεκτικό συνέδριο της Ιταλίας, την δεχότανε και την διαβίβαζε στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Επομένως, η κυβέρνηση προέβη σε μία όχι πολιτική αλλά τεχνική ουσιαστικά διαδικασία διορισμού που φυσικά την ε, διαβίβασε βάσει των συνθηκών. και προέρχεται από τον ανώτατο φορέα, ε, ε, ελεκτικό φορέα της Ιταλίας. Για το τελευταίο ερώτημα τώρα το οποίο μου θέσατε. για το αν θα πρέπει να αποσύρω την υποψηφιότητά μου δηλαδή ή όχι. Εγώ ανέφερα ότι θα πρέπει να ζητήσω την άποψη της κυβέρνησής μου, γιατί στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, όταν πρόκειται μια, για μια θεσμική και όχι ατομική υποψηφιότητα, μου φαίνεται λογικό η κυβέρνηση να μπορέσουν να παρεμβούν στο θέμα αυτό. Η προσωπική μου θέση όμως σε αυτή την περίπτωση θα ήταν προφανώς ότι δεν θα μπορούσα πια να είμαι υποψήφιο, γιατί δεν θα είχα την πλήρη ε, εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι απαράγραπτη για ένα μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Να τελειώσω. Για τον έλεγχο, για το λογιστικό έλεγχο που αναφέρατε, Πρόκειται για ένα έλεγχο χρηστής διαχείρισης και όχι νομιμότητας. Όταν λοιπόν έχει κανείς να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σε σχέση με αυτόν τον έλεγχο είναι κάπως δύσκολο. Εγώ έκανα κάποιες ε, παρατηρήσεις σε σχέση με τη συνέχεια που έπρεπε να δοθεί στο μνημόνιο κατανόησης που είχε κάνει το Υπουργείο το ελεκτικό συνέδριο της, ε, μάλλον το Ιταλικό Υπουργείο σε σχέση με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας για την υπόθεση αυτή των αεροσκαφών. Πιστεύω όμως ότι επί τη βάση αυτών των παρατηρήσεών μου θα υπάρξει εξοικονόμηση χρημάτων για το μέλλον. Δεν ήταν κάτι που αφορούσε μονάχα αυτήν τη συγκεκριμένη απόφαση ενοικίασης. Για το τελευταίο σας ερώτημα, η σχέση μεταξύ του Εθνικού Ελεκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου είναι ζωτική. Γιατί ξέρετε ότι πάνω από 80% των ευρωπαϊκών κονδυλίων τη χάνουν διαχείριση από το κοινό σύστημα και αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων είναι κεφαλαίωδης. Τώρα, οι κανόνες είναι ήδη καταγεγραμμένοι στη συνθήκη στο άρθρο 287 αλλά και στο δημοσιονομικό κανονισμό τη νέα μορφή που έχει τροποποιηθεί το 2006 το άρθρο 53 αναφέρει τη διαδικασία αναφορά ε, απαλλαγής και το γεγονός ότι ο αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει να παρουσιάσει και ένα κατάλογο σε σχέση κατάλογο εθνικών δηλώσεων για τη διαχείριση των κονδυλίων και το Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα η Επιτροπή σας, θα πρέπει να εστιάσεις τις πληροφορίες αυτές. Και με τον τρόπο αυτό το Κοινοβούλιο μπορεί να εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της συνεργασίας. Τέσσερις θέλουν να λάβουν το λόγο. Θέλει κάποιος άλλος να θέσει ένα ερώτημα. Όχι. Προτείνω ο καθένα από τις τέσσερι να θέσει ένα ερώτημα που να μην κρατάει παραπάνω από δύο λεπτά. Και μετά ο κύριο Ρούσο μπορεί να απαντήσει. Ο κύριο Ριβερίνη έχει για δύο λεπτά το λόγο. Ε, it's to you. Ό,τι Συμφωνήστε μεταξύ σας. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς είμαι Ιταλός, αεκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο ε, εξήγησε ο κύριος Ρούσο το γεγονός ότι στην Ιταλία το ελεγκτικό συνέδριο είναι ανεξάρτητο από την πολιτική. Και μάλιστα ακόμα και αυτοί που προτείνουν είναι αποσυνδεδεμένοι από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ακόμα και αν η κυβέρνηση είναι αυτή που προτείνει το όνομα, πάντως ανεξάρτητα γίνεται η επιλογή. Ε, τώρα, πέρα από αυτή την επιτυχία, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού έχει ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των ετών παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν γίνει, φαίνεται απαραίτητο να ενεργήσουμε ώστε αυτού του είδους οι συνεργασίες να γίνουν πιο... η συνεργασία μάλλον να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Με ποιο τρόπο θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο, κύριε Ρούσο. Σας ευχαριστώ. Ας ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε συνολικά. Κύριε Ριβελίνη, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από, τον κύριο Ρούσο τι πιστεύει ότι μπορεί να βελτιώσει την συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το Κοινοβούλιο, γιατί εδώ στην Ευρώπη το ελεγκτικό συνέδριο είναι στην υπηρεσία του ίδιου του Κοινοβουλίου, ακόμα και αν έχει τη δική του ανεξαρτησία. Και πώς μπορείτε τι έχετε σκεφτεί μάλλον για να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα και ποιες είναι οι μεθοδολογίες που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τη συνεργασία. Και επιπλέον σας ρωτώ, πολύ συχνά ε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ε, αναλαμβάνει, μάλλον δέχεται και τις εκθέσεις των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων που πρέπει να εξασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση των ε, ταμείων. Κατά τη γνώμη σας, μια μεταρρύθμιση που να εφαρμόζει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά, προβλέποντας ε, με βάση αυτό το γαλλικό και το βρετανικό ε, ε, ε, μοντέλο όπου το, συνέδριο, το ελεκτικό συνέδριο έχει και δικαιοδοσία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο και έπειτα. Ποιες ιδέες έχετε για να είναι πιο αποτελεσματικό το ελεκτικό συνέδριο. Έχετε κάτι να μας, κάποια ιδέα να μας προτείνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είναι ε, εντυπωσιακές οι γλωσσικές σας ικανότητες και σας ικανότητες. Ε, διάβασα ότι μιλάτε και γερμανικά. Εξού και χρησιμοποιώ τη μετρική μου γλώσσα. Η Ιταλία αποτελεί πηγή πολλαπλών απογοητεύσεων. Ιδιαίτερα εδώ στον έλεγχο προπολογισμού. Εδώ και 10 χρόνια, το συζητήσαμε σήμερα το πρωί και με τον Ισπανό υποψήφιο, εδώ και 10 χρόνια η Ισπανία είναι στην κορυφή των ατασταλιών σε ό,τι αφορά τα διεθντικά ταμεία και αμέσως μετά έρχεται η Ιταλία. 25 ε, υπηρεσίε ελέγχου έχει η Ιταλία και αυτό είναι τμήμα του προβλήματο. Δεν είναι τμήμα τη λύση του προβλήματο. Έχουμε πάρα πολλού εταίρου, πάρα πολλέ ε, ομόλογου και είναι μεγάλο το πρόβλημα να καταλάβουμε ποιο είναι αρμόδιο γιατί, από πού προέρχεται. Um Τι κάνουμε λοιπόν για να βοηθήσουμε τις ε, Ιταλικές αρχές προκειμένου να τα επεξέλθουν καλύτερα σε ό,τι αφορά τις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τι συμβουλή θα μας δίνατε και πώς θεωρείτε ότι θα διαμορφωθεί ο δικός σας ο ρόλος, γιατί θα ήθελα να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος και τώρα ο κ. Σόντεγκάρτεν, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημείωσα την μακρά σας εμπειρία σε ό,τι αφορά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήσασταν επικεφαλής του ελεγκτικού συνεδρίου της Ιταλίας επί 10 χρόνια και ασχοληθήκατε με τέτοια θέματα ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέματα απάτης επίσης με τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία θα μπορούσατε να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση για το ποια θεωρείτε ότι είναι τα δύο-τρία μεγαλύτερα προβλήματα. Ποιες χώρες είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά ταμεία. Και να μας πείτε κατά πόσον εκτιμάτε ότι έχει σημειωθεί η βελτίωση και κατά πόσον θεωρείτε ότι η Ιταλική κυβέρνηση εργαζόταν προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας βελτίωσης. Αυτά φυσικά ε, για την περίοδο κατά την οποία εργαζόσασταν για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούσο. Έχετε περίπου πέντε λεπτά αν θα θέλετε να απαντήσετε λίγο ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Ακόμη και αν καταλαβαίνω πως δεν είναι εύκολο να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα θέματα που είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα και να τα αναφέρουμε όλα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό θα απαντήσω από κοινού για να μπορέσω να συνδυάσω τα ερωτήματα που έχουν κοινά στοιχεία. όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του, μάλλον μεταξύ του Ελληνικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα όσα ήδη είχα πει απαντώντας στην ερώτηση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ο Ευρωπαίος ε, νομοθέτης το έχει συνειδητοποιήσει εξ αρχής. Είναι σαφές ότι το ελεγκτικό συνέδριο ως εξωτερικός ελεγκτής ε, δημιουργείται ταυτόχρονα με τη φάση όπου το Ευρωκοινοβούλιο αποκτά εξουσίες όσον αφορά τον προπολογισμό και χρειάζεται για την δική του πολιτική κρίση για την ε, διαχείριση από πλευρά της Κομισιόν τη στήριξη ενός τεχνικού οργάνου. Άρα λοιπόν οι σχέσεις μεταξύ των δύο οργάνων είναι ε, διάρρηκτες και ε, το σύστημα ήδη νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και βασίζεται στην διαδικασία απαλλαγή. Μπορεί να Υπάρχει ήδη ένας ε, ενάρετος κύκλος, θα έλεγα εγώ, input και feedback ανάμεσα στα δύο όργανα και συγκεκριμένα αυτήν εδώ την Επιτροπή, διότι το ελεγκτικό συνέδριο εντοπίζει τους κινδύνους στη διαχείριση του προπολογισμού και τους εντοπίζει στις εκθέσεις του. Κάνει τους ελέγχους του, φτιάχνει τις συντάσεις της εκθέσεις του το το, και τα υποβάλλει στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο λοιπόν αξιολογεί αυτές τις εκθέσεις και προβαίνει στις απαλλαγές ή όχι και στρέφεται ξανά στο ελεγκτικό συνέδριο για περαιτέρω ελέγχους. Είναι προνομιακή η σχέση γιατί υπάρχει μια διαρκή συνεχιζόμενη ε, σχέση μέσα στην ίδια χρήση κάθε φορά. Και τώρα υπάρχει και ενίσχυση, θα έπρεπε να, μάλλον, να ενισχυθεί περισσότερο η πτυχή που σχετίζεται με το άρθρο 319 μέσω του οποίου η Επιτροπή οφείλει να εκτελεί τις συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για έτσι έτσι ώστε το, το ελεγκτικό συνέδριο να έχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια και να ξεκινήσει ένα νέο γύρο ελέγχων. Και από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τη δευτερογενή ε, νομοθεσία, στον δημοσιονομικό κανονισμό υπάρχει η αρχή σύμφωνα με την οποία η Κομισιόν οφείλει να υποβάλει ένα κατάλογο ετήσιο των ελέγχων για την νομιμότητα και την ε, συμμόρφωση που γίνεται σε εθνικό επίπεδο για τις πληρωμές και τις πιστοποιήσεις και από εκεί μπορεί να ξεκινήσει το συνέδριο αν το κοινοβούλιο κάνει ε, παρατηρήσεις για να κάνει τους ελέγχους του. Και αυτό το συνδέω με την τελευταία φάση, τις σχέσεις δηλαδή του ελεγκτικού συνεδρίου με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, γιατί κατά τη γνώμη μου Όλα αυτά σημαίνουν πως τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, εφόσον ελέγχουν αυτές τις πτυχές νομιμότητας των πληρωμών από πλευράς των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων, μάλλον των εθνικών αρχών, θα συμμετέχουν περισσότερο σε όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό συνδέεται και με τις εθνικές δηλώσεις, γιατί έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να το λάβει υπόψη και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα έχει feedback. Όσον αφορά τη δομή, πιστεύω πως αυτή τη στιγμή το ελληνικό συνέδριο είναι αποτελεσματικό και μπορέσαμε να φτάσουμε σε μια καλή συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην απέτηση για την ε, ταχύτητα των ε, αποφάσεων και επιπλέον είναι έχουμε από την άλλη πλευρά την άλλη απέτηση ώστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κάθε κράτος έχει τις δικές του παραδόσεις, ιστορία και ήθη και έθιμα να μπορεί να κάνει τη δική του συμβολή. Στην κυρία Γκρέσλε, θέλω να την ευχαριστήσω για τις πολλές ε, ερωτήσεις της. Δυστυχώς στα Ιταλικά μονάχα θα μπορέσω να τις απαντήσω. Δεν είμαι σε θέση να μπω σε λεπτομέρειες, δεν θα είχαμε και το χρόνο όσον αφορά τις αρχές τις ελεγκτικές αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Πιθανότατα θα είναι πολύ άριθμες. Η Ιταλία ανέκαθεν ναι, έχει την τάση να φτιάχνει ένα σωρό ωραιότατους κανονισμούς που όμως στην συνέχεια δεν φαίνεται να είναι εύκολα εφαρμόσιμη. Πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται στην αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού που αναφέρεται και που αφορά τις δηλώσεις αξιοπιστίας που εκδίδουν οι ελεγκτικές αρχές σε εθνικό επίπεδο. Και έτσι θα μπορούσε να εμβαθυνθεί ο έλεγχος με δυνατότητες βελτίωσης σύντομα της κατάστασης τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο δικαστήριο και στα... Συγγνώμη, όχι το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια με τη σειρά τους. Τώρα, για τις απάτες. Εγώ ασχολήθηκα με τη δημιουργία της ε, Ούκλαφ και μετά της Όλαφ και γνωρίζω τη σοβαρότητα του προβλήματος ως εκ τούτου. Θα πρέπει να πούμε πως εν γέννη ο ρόλος του ελεγκτή δεν μπορεί να είναι θεσμικά ο ρόλος του ερευνητή ή του αστυνομικού δεν έχει το δυνατό, τη δυνατότητα να κάνει τέτοιου είδου έρευνε, ε, ένα ε, εκπρόσωπο του συνεδρίου ούτε και μπορεί άμεσα να παρέμβει για να καταστήλει ο ρόλος μας περισσότερο συνίσταται στην πρόληψη, να εντοπίσουμε δηλαδή τους τομείς κινδύνου και τις μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να οδηγούν σε υποψίες για απάτη και με τους ελέγχους σωστής διαχείρισης, εντοπίζοντας τις αδυναμίες των συστημάτων διαχείρισης και κάνοντας συγκεκριμένες συστάσεις ώστε να βελτιωθούν τα συστήματα και να ενεργήσουμε έτσι με αποτελεσματικό, πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Εγώ, αν διοριστό μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η προσοχή μου θα είναι στραμμένη σε αυτό το πρόβλημα και ελπίζω ότι η εμπειρία μου θα είναι χρήσιμη. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρούσο. Ως ήθεστε, η εισηγήτρια θα συνοψίσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούσο για τις απαντήσεις του και φυσικά τους συναδέλφους μας να τους ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις τους που μας βοήθησαν να καταλάβουμε πολύ καλύτερα μεταξύ άλλων και το Ιταλικό σύστημα για την ε, πρόταση υποψηφίου στο Ελληνικό συνέδριο που αφαιρεί βέβαια τις πολιτικές ε, ε, σκοπιμότητες σε ό,τι αφορά το διορισμό κάποιου υποψηφίου. Ίσως θα πρέπει να το λάβω υπόψη και στον επόμενο κανονισμό για διορισμό στο ελεκτικό συνέδριο. Μπορεί να είναι πολύ θετικό αυτό ο μηχανισμό. Κατά τα άλλα, σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι ξέρουμε πολλά ήδη πράγματα, αρκετά για να μπορέσουμε να πάρουμε μια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλο των ακροάσεων των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Σα ευχαριστώ κύριε Ρώση, λέει Και τώρα διακόπτουμε για λίγα λεπτά και θα συνεχίσουμε σε κεκλεισμένων το θυρών τη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν λειτουργικότητα σε ό,τι αφορά την παρουσία τους να αποχωρήσουν.